Uh, uh, Σα ενημερώνω ότι έχω λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ειδοποίηση για την εκλογή της κυρίας Μπομπέτ ε, Βίντερ ε, και θα αντικαταστήσει τον κύριο Γιάκομ και ανατρέχει η αντικατάσταση της 10 πρώτου του 19. Καλώς όρισε η συνάδελφος και υπενθυμίζω ότι θα είναι τακτικό μέλος του Κοινοβουλίου και στα όργανα αυτού έχοντας ε, όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον κανονισμό. Και πάλι καλώς όρισε. Όπως έλεγα, συνεχίζονται οι εργασίες της Σύνοδο. Έχουμε τα χθεσινά πρακτικά τα οποία είναι διαθέσιμα για όποιον θέλει. Έχετε κάποιο σχόλιο για τα πρακτικά. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως εγκρίνονται. Και πάμε στο επόμενο θέμα της Μεσσίας Διατάξεως που είναι τα επίκαιρα θέματα του άρθρου 153 του Α του κανονισμού. Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος. Σας ενημερώνω ότι δεν προβλέπεται κάτι για αυτή τη συζήτηση, ούτε μπλε κάρτες. Οπότε, παρακαλώ, τώρα για λογιασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να λάβει τον λόγο κύριος Κόβατσος. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχουμε 30 χρόνια από τότε που κατέπεσε το Κομμουνιστικό Καθεστώ Ανατολική Ευρώπη και πριν από 10 χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε αυτό το ψήφισμα όσον αφορά την συνειδητοποίηση ε, της Ευρωπαϊκής ε, Μνήμης για τον ολοκληρωτισμό. Πρόκειται για καταδίκη όλων των ολοκληρών καθεστώτων των 20ου αιώνα. Οπότε ε, θα πρέπει να εξισώσουμε κατά κάποιο τρόπο τον φασισμό, τον ναζισμό με τον κομμουνισμό και τα όσα δεινά προκάλεσαν. Αν αντλήσουμε κάποια μαθήματα από τα τραγικά αυτά γεγονότα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα θωρακίσουμε την δημοκρατία. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή ενότητα κράτος δικαίου, σεβασμό ελευθερίας και αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουμε, να φρενάρουμε το μίσος, την ξενοφοβία, τις ολοκληρωτικές ιδέες, να μην φουσκώνει το ποτάμι του στην κοινωνία μας και είχαμε πει ότι θα, έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτή η ζήτηση, αλλά δεν έγινε ποτέ έχουμε ένα σωρό προκλήσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιδράσαμε, αντιδράσαμε ε, και ε, θα έπρεπε να έχουν προλιάνει το έδαφος για αυτή την ε, ε πέτειο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα, τα φαντάσματα του παρελθόντος. Μα οι εθνικισμοί τώρα έχουν φουντώσει. Θα πρέπει να θυμόμαστε, θα πρέπει να καταλάβουμε την ιστορία μας και τι πάει να πει ολοκληρωτικό καθεστώς αρκεί να ρίξουμε μια ιστορία συγκεκριμένων χωρών. Εκεί οι νέοι έχουν απογοητευτεί, δεν έχουν οικονομικές προοπτικές, δεν υπάρχει ισότητα και έχουν στραφεί προς άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. αυτό αρκεί για να μας πείσει για το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος επανάληψης των σφαλμάτων του παρελθόντος. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μνήμη, ιστορική μνήμη. Είναι να μην είναι στόχοι ε, αυτών των κομμάτων που προσφέρουν τις εύκολες λύσεις. Αν δεν θυμόμαστε το παρελθόν, τότε αφήνουμε το περιθώριο να παραπλανηθούν οι νέοι, να υπάρχει παραπληροφόρηση για, από πλευράς φασισμού, ναζισμού και κομμουνισμού. Αυτοί εκμεταλλεύονται την νοσταλγία που υπάρχει σήμερα γιατί υπάρχει άγνοια σχετικά με τα εγκλήματα αυτών των ιδεολογιών και σε κάποιες χώρες λοιπόν υπάρχει νοσταλία για τον σταλινισμό, υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές και βέβαια θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει ένα μοντέλο που να βοηθήσει. Παντού, παιδεία. Παιδεία για την επόμενη γενιά Ευρωπαίων. Για όλη την Ευρώπη. Να μάθουν τι θα πει ολοκληρωτικό καθεστώς. Να μάθουν το πόσοι θυσιάστηκαν για ελευθερία και δικαιώματα. Δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η ελευθερία. Όπως έλεγε κάποιος φιλόσοφος, είναι μια γενιά μακριά το σβήσιμο της φλόγας της ελευθερίας. Έχουμε την 20η περίοδο του ευρώ, αλλά δεν είναι το ευρώ η Ευρώπη. Όχι, δεν είναι μόνο η ενιαία αγορά θα πρέπει να έχουμε εγγύσεις για δικαιώματα και ελευθερίες. Η Ένωση είναι απάντηση στη φρίκη του ολοκληρωτισμού. Το τίμημα ήταν εκατομμύρια αθώων θυμάτων. Μεγάλο βάσανο για όλους. Οπότε να συνειδητοποιήσουμε ότι η απειλή έγκυται στην έλλειψη ιστορικής μνήμης. Με την παιδεία να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα της μνήμης για την επόμενη γενιά, να μην γίνει η επόμενη γενιά θύμα χειραγώγησης λόγω της άγνοιας. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το θέμα που συζητάμε σήμερα βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη τον τελευταίο αιώνα παραμένουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις κοινέ αξίες και στις γενικές αρχές του σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στόχος είναι να προωθήσει αυτές τις αξίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν πολλές οι προκλήσεις και πολλές οι δυσκολίες για αυτές τις αξίες τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς οι νέες γενιές δεν έχουν υποφέρει κάτω από απολυταρχικά καθεστώτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμη ε, ο κίνδυνος να θεωρήσουν δεδομένες αυτές τις κοινέ αξίες. Οι κοινέ μας αξίες ε, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε την μακρύτερη περίοδο ειρήνης στην Ευρώπη. Παραμένουν ακρογωνιαίος λήθος για τη δημοκρατική μας κοινωνία και θα πρέπει συνεχώς να τις καλλιεργούμε. Σήμερα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ανοιχτή μας κοινωνία, είτε μέσω της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, των διακριτικών μεταχειρήσεων ή του ρίζοσπαστισμού και της βίας. Κατανοώντας το παρόν και για να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν, χρειάζεται να γνωρίζουμε καλύτερα το παρελθόν. Γνώση για τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητες για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Με τη γνώση, δεν θα, ε, με τη γνώση του παρελθόντος, οι πολίτες ε, θα έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν ε, τη δική τους γνώμη για την τρέχουσα ιστορία. Παράλληλα, προωθείται ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση και η συνεργασία που ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι η παιδεία παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των κοινών μας αξιών και στην προώθηση της κοινή κατανόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, των άλλων πολιτών. Όλοι γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της εκπαίδευσης είναι περιορισμένη και τα κράτη-μέλη παραμένουν απολύτως υπεύθυνα για το εκπαιδευτικό του σύστημα και για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Παρ' όλα αυτά, σε μια εποχή που η Ευρώπη κοιτάζει προς το μέλλον και προσπαθεί να ε, ξαναφέρει κοντά τους πολίτες και ιδίως τους νέους γύρω από ένα θεματολόγιο κοινών αξιών, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ των Ευρωπαίων. Υπό αυτή την έννοια, τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις οι οποίες εκδηλώνονται με διάφορες πολιτικές δηλώσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις του Συμβουλίου που αποτελούν τη βάση για συνεργασία σε αυτό τον τομέα. Στη διάσκεψη κορυφής του Γκέτεμπουργκ τον Νοέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν την παιδεία και τον πολιτισμό ως το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί στην ημερήσια διάταξη των ηγετών σε αυτούς τους τομείς. Η συζήτηση στο Γκέτεμπουργκ ε, ε, ακολουθήθηκε από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2017 που τονίζουν τη σημασία του πολιτισμού και της παιδείας για τη δημιουργία μιας κοινωνίας συνοχής. Τον Μάιο του 2018 το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα προωθώντας τις κοινέ αξίες και την πολυσυλλεκτική εκπαίδευση. Αυτή η σύσταση ακολουθούσε την δήλωση του Παρισιού του 2015, στην οποία οι Υπουργοί Παιδείας τονίζουν τη σημασία του ρόλου της εκπαίδευσης. Οι δεσμεύσεις της δήλωσης του Παρισιού έχουν και σήμερα την ίδια σημασία όπως και τότε και είναι εξίσου επίκαιρες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το Erasmus Plus, το Horizon, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, όλες τις πρωτοβουλίες που θα υποστηρίξουν τις κοινέ μας αξίες πρέπει να δώσουμε στους νέους μας τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι υπεύθυνοι πολίτες με σωστή ενημέρωση. Η κριτική σκέψη αποτελεί βασικό στοιχείο για την κοινωνία του σήμερα. Οι νέοι μας πρέπει να αναπτύξουν τη δυνατότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης για να αντιμετωπίζουν τον αυξανόμενο όγκο πληροφόρησης πρέπει να έχουν επίγνωση της ανάγκης να αναγνωρίζουν ε, τις αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και να αναγνωρίζουν και τον κίνδυνο παραπληροφόρησης. Και τέλος, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενθαρρύνουμε ε, την ε, ανεκτικότητα και τον αμοιβαίο διάλογο για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον βασικό ρόλο παίζει και η συνεχής ανάπτυξη των νέων και του προσωπικού γενικότερα. Είναι σημαντικό να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ευαίσθητα θέματα ή αντιφατικά ζητήματα και να μην αφήνουμε αναπάντητες τέτοιες ερωτήσεις. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι διδάσκοντες θα πρέπει να υποστηρίζονται στην δύσκολη δουλειά τους ε, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Το θέμα αυτό συνδέεται στενά με τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας όπως παρουσιάστηκαν χθε από τον Πρωθυπουργό. Ένας από τους βασικούς κανόνες ε, είναι ο πυλώνα ε, των ευρωπαϊκών αξιών. Πρέπει να τονίσουμε την αλληλεγγύη και τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντα πολιτικές ε, που καταπολεμούν τη διακριτική μεταχείριση, που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση και επίσης αυξάνουμε τη συμμετοχή των πολιτών και ιδίως των νέων στις ε, συζητήσεις για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα αυτό θα παραμένει υψηλή προτεραιότητα στο πολιτικό θεματολόγιο του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία ε, Υφυπουργέ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο, Γιούροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προβλέψατε αυτή την τόσο σημαντική και ιδιαίτερα επίκαιρη συζήτηση. Το να μάθει κανεί για την ιστορία μα και να αναλύσει τι ε, περίπλοκε δυνάμει ε, οι οποίε αναπτύσσονται στι κοινωνίε μα, αυτό είναι η βάση για να κατανοήσει κανεί τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Το να γνωρίζουμε το παρελθόν μας είναι καθοριστική σημασία για τη δημιουργία του μέλλοντος της Υπήρου μας και των χωρών μας. Να μην ξεχνάμε ότι οι ιδέες που χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, Ολοκλήρωσης βασίζονται στο ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η σκοτεινή ε, πλευρά της ιστορίας και πρέπει να υπερασπιζόμεθα αυτή την άποψη κάθε μέρα το να ε, θυμόμαστε ε, και να διδάσκουμε το παρελθόν, όπως επίσης και το να καλλιεργούμε τη μνήμη σε πολυτάραχες εποχές, αυτό είναι ένα κλειδί για το κοινό μας μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να περιλαμβάνονται στην πολιτική μας, ε, όπως κάνουμε και με το να υπάρχει ε, μία ε, ημέρα για να θυμόμαστε αυτά τα καθεστώτα. Είναι 23η Ιουνίου κάθε χρόνο. Εμείς στηρίζουμε την έρευνα σε θέματα ολοκληρωτισμού, το να διαφυλάσσουμε τη μνήμη του ολοκληρωτικού καθεστώτος της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα από τα κομβικά θέματα του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες. Ένα πρόγραμμα που στηρίζει δραστηριότητες ε, που έχουν σχέση με την πολιτιστική ε, ποικιλομορφία και τις ε, πολιτιστικές αξίες. Υπάρχουν κονδύλια για να αντιμετωπίσει κανείς την, τα απολυταρχικά καθιστώτα στην Ευρώπη και για να ε, θυμούμαστε τα θύματα. Επιπλέον η Ευρώπη για τους πολίτες ε, είναι το βασικό εργαλείο της Ευρώπης για να στηρίξει πρωτοβουλίες ε, που ευαισθητοποιούν και εκπαιδεύουν σχετικά με το ολοκαύτωμα. Κάθε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν ε, διάφορες διαδηλώσεις σε μνήμη σχετικά με το ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητά μας. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έχει ε, αποκτήσει την θέση του μόνιμου ε, κράτους μέλους στην συμφωνία και στη συμμαχία που υπάρχει για το ολοκαύτωμα. Είναι σημαντικό το ότι διαθέτουμε 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα σε σχέση με το ολοκαύτωμα. Επιπλέον, Όσον αφορά την έρευνα, το 2015 και το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 ε, στηρίζει ε, την αντίδραση στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες έτσι ώστε να υπάρχει αλλοκατανόηση στους Ευρωπαίους μέσα από τη δουλειά για το πολιτάραχο παρελθόν. Έχουμε το crash το οποίο εκπροσωπεί την πολιτιστική αντίσταση στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει δημιουργήσει την πρώτη ψηφιακή τράπεζα δεδομένων και προβάλλει τις πρώτες μορφές πολιτιστικής αντίστασης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Ε, στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι αυτά τα στοιχεία, τα πολιτιστικά, είναι καθοριστική σημασία έτσι ώστε να υπάρχουν πλουραλιστικές δημοκρατίες. Στον τομέα της εκπαίδευση η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει εθνικές πολιτικές με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας μας και των κοινών μας αξιών. Το νυν πρόγραμμα Erasmus ΣΥΝ έχει στηρίξει περίπου 30 προγράμματα που ασχολούνται με την ιστορία και τον ολοκληρωτισμό στην Ευρώπη. Τα προγράμματα αυτά έδωσαν την ευκαιρία στους πολίτες και στους φοιτητές να μάθουν για το παρελθόν με άμεσο τρόπο και να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους ε, ως ένα ευκταίο αποτέλεσμα. Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σύσταση του Συμβουλίου για την προαγωγή κοινών εξιών, συμπεριλαμβανομένης και της παιδείας ε, και της διδασκαλίας. Τα κρατημέλη συμφώνησαν από αυτού μετά από κάποιους ε, μήνες και αυτό ήταν ένα πραγματικό ορόσημο. Ποτέ κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε πει με τόσο μεγάλη σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι να προαχθούν οι κοινέ αξίες μας, να υπάρχει η αίσθηση του ότι όλοι ανήκουμε σε ένα κοινό ε, πλαίσιο και το πιο σημαντικό από όλα να μάθει κανείς για τις περίπλοκες πολιτιστικές και άλλες εμπειρίες στα κράτη-μέλη μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι η ε, παιδεία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να ε, προλάβουμε τον αντισημιτισμό και γι' αυτό η Επιτροπή χρηματοδοτεί μία μελέτη που φέρει τον τίτλο «Το ολοκαύτωμα σε σύγχρονες ε, μορφές εκπαίδευσης». Μαζί με την UNESCO γίνεται αυτό. Και τέλος μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε καλύτερα για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και είμαι υπερήφανη που η ετικέτα Ευρωπαϊκή Κληρονομιά έχει ε, αποδοθεί σε σημαντικούς χώρους που υπάρχουν ε, μεταξύ άλλων στα ναυπηγεία Ντάνσκα της Πολωνίας ή στο μνημείο Σίκαρτ στην ε, Ρουμανία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να προβάλλει τη μνήμη του σε απολυταρχικά καθεστώτα, ανεξάρτητα με το ποια είναι η ιδεολογική τους βάση. Να κατανοήσουμε τον παρελθόν μας είναι καθοριστική σημασία αν θέλουμε να ζήσουμε μαζί και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ήπειρό μας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, είναι πολλοί αυτοί που έχουν γραφτεί για να λάβουν το λόγο. Θα κρατήσει πολύ η συζήτηση αυτοί και άλλες. Οπότε, σεβαστείτε τα χρονικά όρια αγορεύση. Δύο λεπτά η κυρία Καλνίδα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κατά τον τελευταίο αιώνα διδαχθήκαμε ένα μήνυμα σκληρό. Πώς δικτατορίες είναι αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα εγκλήματά τους. Παιδεία, έρευνα και μνήμη. Έτσι θα είμαστε ανθεκτικοί, θωρακισμένοι εναντί αυτών. Να έχουμε λύσεις δημοκρατικές στις κοινωνίες μας. Αναγνώριση και αντίσταση προς ριζοσπάστες, λαϊκιστές, ακραίους δεξιάς και αριστεράς. Να μην τους αφήνουμε να αμαυρώνουν τις μοναδικές αξίες, να μην ε, κάνουν πλήση εγκεφάλου στην κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε μετά το τραύμα που είχαμε από τον εθνικό σοσιαλισμό και τον ε, κομμουνισμό και έχουμε όλους αυτούς τους λαϊκιστές χειραγωγούν για να αποκτήσουν την εξουσία και να στήσουν σκληρά καθεστώτα εις βάρος εκατομμυρίων. Τι λέει η ιστορική εμπειρία στη Δυτική Ευρώπη. Ήταν ο ναζισμός. Σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαμε και ναζισμό και κομμουνισμό και τους δύο. Πρόκειται για ολοκληρωτικά καθεστώτα που είναι τώρα η κοινή μας κληρονομιά και άρα θα πρέπει με μία γλώσσα η Ευρώπη να αποφανθεί για αυτό το ιστορικό κληροδότημα, να έχουμε ένα πλαίσιο, να έχουμε πρικοδότηση αρκετή για να γίνει ιστορική έρευνα και όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσον αφορά κάθε πρόγραμμα σχετικό, θα πρέπει να μπορέσουμε να ψάξουμε τα ιστορικά μας αρχεία, να δούμε τι ιστορικά ψέματα έχουν εξυφανθεί και να δούμε τη σχέση μεταξύ λαϊκισμού, εξτρεμισμού, ε, αυταρχισμού για όλο τον κόσμο επίσης θα πρέπει να ενεργήσουμε ε, κάτι να κάνουμε για παραβίαση των δικαιωμάτων σε Ιράν, Κίνα, Ρωσία ή από τους τζιγαντιστές. Και σταματάει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την κυρία Κάμερφερτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρώπη, ειδικά τον 20ο αιώνα, παρουσιάζει μια ιστορία των παραπλανήσεων, των εγκλημάτων, του πολέμου, των αδικιών, αλλά και μια ιστορία των επιτυχιών. Έχουμε την σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και την περίπτωση της άρσης του σιδηρού παραπετάσματος και της εμβάθυνση ε, τη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η δημοκρατία χρειάζεται τη μνήμη. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μέλλον. Η σύσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή υπεράσπιση των βασικών αξιών είναι ένα μάθημα που μαθαίνουμε από το πιο σκοτεινό κεφάλαιο τη ιστορία του 20ου αιώνα το βλέμμα στο παρελθόν, βοηθάει να έχουμε λύσεις για το μέλλον, αναγνωρίζοντας τα λάθη, συνειδητοποιώντας πώς φτάσαμε στα λάθη αυτά και βεβαίως αναγνωρίζοντας και την ευθύνη, ακόμα και για πράξεις για τις οποίες κανείς δεν ήταν υπέτειος. Ε, το να πέσει στα γόνα το Βίλι Μπραν στη Βαρσοβία, αυτό είναι το καλύτερο δείγμα το ότι πολλοί δέχτηκαν την ευθύνη τους. Βέβαια, θέλω να σας προειδοποιήσω, όχι με αυτά να κάνουμε πολιτική, αυτό δεν γίνεται. Η ιστορία είναι πάντα μακρά, περίπλοκη, αντιφατική ακόμα και στην ίδια της ε, την ε, αφήγηση. Ε, δεν υπάρχει μία και μόνη αλήθεια. Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που δεν μπορεί κανείς να τα παρνηθεί, αλλά από την άλλη το να θυμόμαστε πράγματα, ε, να λέμε ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις και ότι υπάρχει μία και μόνο άποψη, αυτό είναι ανόητο. Και αυτό δεν ενώνει, αλλά διχάζει. Το να θυμόμαστε πράγματα, αυτό βοηθάει μόνο αν θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο μανιχαϊσμός, άσπρο-μαύρο, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ε, το να απαντήσει κανεί την επαιτειότητα και την αθότητα αυτό δεν είναι απλό. Το να θυμόμαστε πράγματα αυτό βοηθάει αν νιώθει κανείς και κάποιες αμφιβολίες. Και γι' αυτό βοηθάει αυτή η τάση και έναντι του λαϊκισμού. Μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τα όρια μας. 30 χρόνια μετά την άρση του σιδηρού παραπετάσματος θα πρέπει να γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε ότι εκείνοι που τότε θεωρούσαν ότι έχει την μία και απόλυτη αλήθεια, αυτοί ανατράπηκαν. Ο ολοκληρωτισμός ε, και ο αυταρχισμός έχουν ένα πράγμα κοινό. Δεν λένε να θυμόμαστε, αλλά αφηγούνται ιστορίες και νομίζω ότι αυτή τη διαφοροποίηση θα πρέπει να τη γνωρίζουμε. Να τα πούμε αυτά στα παιδιά μας για να είναι θωρακισμένα. Ευχαριστώ πολύ. θα πρέπει να τηρούμε το χρόνο για να σεβόμαστε και το χρόνο των άλλων συναδέλφων. Θα είμαι αυστηρός λοιπόν με την τήρηση του χρόνου. Έκανα ήδη δύο σφάλματα, σα άφησα να μιλήσετε περισσότερο, αλλά θα είμαι αυστηρό στο εξή. Επόμενος ομιλητής, Σκρίπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Πολλοί βουλευτές έχουν νιώσει στο πετσί τους το τι σημαίνει αυταρχικό καθεστώς που επί 40 χρόνια σε πολλά κομμάτια της Ευρώπης τους έκανε να υποφέρουν. Εγώ είμαι ένα παιδί από ένα τέτοιο καθεστώς. Ήμουν σε οργανώσεις νέων, ήμουν υποχρεωμένος να υπερασπιστώ τη χώρα μου, αλλά μας είχαν ε, πείσει ότι ε, οι θεωρίες του μαρξισμού του Λένιν ήταν ε, οι καλύτερες θεωρίες και ότι η θρησκευτική λατρεία ήταν κάτι το εσφαλμένο. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας μαθαίνοντάς τους αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας για να μην επαναληφθεί ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν η μνήμη να βοηθήσει ένα στρατιώτη, ο Γιώζεφ Γκάπτσικ, που κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν στον στρατό της ε, Τσεχοσλοβακίας και συμμετείχε σε ε, μια συγκεκριμένη επίθεση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους μας για την ύπαρξή του. Γεννήθηκε από τις στάχτες η Ένωση, τις στάχτες αυτών των ε, δικτατοριών, αλλά ήταν έναντι αυτών των αυταρχικών καθεστώτων ένα καταφύγιο. Θυμάμαι τι είπε ο Βάτσλαβ Χάβελ, πρόεδρε. Μας είπε το πόσο μοιάζουν οι ρίζες αυτών των διαφορετικών ολοκληρωτισμών τι γίνεται με αυτές τις ιδεολογίες, το πόσο άσχετες είναι με την πραγματικότητα και με τη ζωή. Γιατί η ιδεολογία υποκαθεστά τη λογική σε αυτά τα καθεστώτα και η αλήθεια ταυτίζεται με την εξουσία. Εάν χαλαρώσουμε την προσοχή μας, εάν δεν θυμόμαστε το παρελθόν, εάν δεν θυμόμαστε την παράδοση της λογικής, ε, το, το, το, το πώς θα ξεπεράσουμε όλες τις διαιρέσεις, τότε τι θα γίνει θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις πρωτοβουλίες για έρευνα, για παιδεία, να μην φτάσουμε σε αυτή την τρέλα του ολοκληρωτισμού. Γιατί το, το λέγανε τυραννία οι αρχαίοι. Ε, χρειάζεται μια πάλι για όλη την Ένωση. Γιατί πρόκειται για κάποια κληροδότημα πολύτιμο η δημοκρατία. Χρειάζεται να την προσέξουμε, να τη φροντίσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη του ολοκληρωτισμού. Αυτό να γίνει μέσα από την προοπτική της ευρωπαϊκής ιστορίας, της κοινή μας ιστορίας και να μην οδηγηθούμε σε εθνικισμούς, να μην ρίξουμε νερό στο μήλο του εθνικισμού και έτσι να τιμήσουμε, να αναδείξουμε την αλήθεια. Υπάρχει μία αλήθεια, υπάρχει κάτι αντικειμενικό και φωτεινό για αυτό που είναι η έμπνευση για όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Ροπέ. Ένα λεπτό. Ναι, είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε κυρίως τους νέους τις τραγωδίες που υπέστη ο κόσμος λόγω των ολοκληρωτισμών. Τι έγινε στην Λιθουανία από την σοβιετική κατοχή. Έχασαν τη ζωή τους περίπου 800.000 συμπατριώτες μας. Τους στείλανε στη Σιβηρία, τους περισσότερους από αυτούς, για να πεινάσουν, να αρρωστήσουν και πέθαναν ε, παιδιά και ενήλικες υπό τρομερές συνθήκες, κομμουνιστικά εγκλήματα που δεν έχουν καταδικαστεί επαρκώς. Οι συνέπειες ζουν ακόμα σήμερα ο σταλινισμός διαφημίζεται στην ε, Ρωσία. Το σοβιετικό καθεστώς αποτελεί κάτι σαν είδωλο σε μαγαζιά με σουβενίρ, σε προγράμματα τηλεόρασης. Ακόμα και η συμφωνία με το Χίτλερ του Στάλιν εις βάρος των Βαλτών είναι κάτι το οποίο διαφημίζεται. Ο επόμενος. Ο κύριος Χουντής, 1,5 λεπτό. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα έχει αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα και τι προκλήσει τη νεολαία και τη εκπαίδευση. στι μέρε μα ο ευαίσθητο κλάδο τη εκπαίδευση με την επίθεση που δέχεται κινδυνεύει να μην μπορεί να επιτελέσει τον ιστορικό και κοινωνικό του ρόλο. οι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ τη ευρωπαϊκή ένωση έχουν οδηγήσει στην αποδιάρθρωση στον κατακαιρματισμό τη εκπαίδευση προτάσσοντα την ιδιωτικοποίηση ω πανάκια με βάση τι επιταγέ τη αγορά οι περικοπέ των δημοσίων δαπανών και η υποχρηματοδότηση έχουν απαξιώσει τα εκπαιδευτικά συστήματα και έχουν υποβαθμίσει την ποιότητά του. η σημερινή συζήτηση συνδέεται άμεσα με αυτή την ποιότητα το περιεχόμενο και τη συμβολή τη εκπαίδευση που στο όνομα όμω τη θεωρία όπω αναπτύχθηκε το δύο άκρων προσπαθεί να αποπροσανατολίσει να ξαναγράψει την ιστορία και να δικαιολογήσει κατά την άποψή μου τα μέτρα που λαμβάνονται σε ορισμένε χώρε κατά των κομμουνιστικών και αριστερών κομμάτων. αγαπητοί συνάδελφοι τι ιστορικό μάθημα δίνει η άρνηση τη γερμανία να αποπληρώσει το κατοχικό δάνειο που πήρε από την ελλάδα να αποπληρώσει και να αποζημιώσει τα θύματα της ναζιστικής κατοχής. ποιο είναι το ιστορικό μάθημα που δίνουμε και η αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης. αγαπητοί συνάδελφοι τούτες τις μέρες τούτες τις ώρες η παιδεία στην ελληνική πραγματικότητα δέχεται μια νέα επίθεση λιτότητας από την κυβέρνηση περικοπής των δαπανών και αλλίωση των πτυχίων αυτοί οι καταστροφικοί σχεδιασμοί δεν εξυπηρετούν τι ανάγκε ούτε τη παιδεία ούτε των κοινωνιών μα. η αγωνιστική στάση σπουδαστών και καθηγητών αυτή την περίοδο που αντιμετωπίζουν αυταρχική βία δείχνει τον δρόμο για μια καθολική εκπαίδευση και εκπαιδευτικού με αξιοπρέπεια και εργασιακά δικαιώματα. σα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Uh, Όσοι δεν διδάσκονται από την ε, ιστορία είναι καταδικασμένοι να επαναλάβουν τα σφάλματα. Πιστεύω στην εκπαίδευση, αλλά ξέρω ότι η εκπαίδευση χρησιμοποιείται για να προωθήσει την προπαγάνδα. Ανησυχώ διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως τρόπο προώθησης ε, ε, της προπαγάνδας της για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσει να μετατρέψει τους πατριώτες πολίτες ε, σε ε, κάποιους οι οποίοι θα είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι θα πει λαϊκιστής. Το αντίθετο του λαϊκιστής είναι αυτός που είναι κατά του λαού, αντιλαϊκιστής οι λαϊκιστές, ε, όπως τους αποκαλείτε, λένε αυτό που δεν θέλετε να ακούσετε και συχνά ε, ανησυχώ με το ψεύδος που επαναλαμβάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αιτία για 25 χρόνια ειρήνη στην Ευρώπη. Πολύ συχνά βοηθάει η επικοινωνία και η μνήμη, αλλά να μην ξεχνάμε και το ρόλο που έπαιξε το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, τα Ηνωμένα Έθνη και, πιστέψτε το, και τα πυρηνικά όπλα. Η απειλή, των πυρηνικών όπλων κατέστησε αδύνατο τον πόλεμο. Αν λοιπόν μιλάτε για την εκπαίδευση, αφήστε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν τι θεωρούν καλύτερο για τα δικά τους παιδιά σε κάθε κράτος μέλος. Δείξτε εμπιστοσύνη στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και αφήστε την πολιτική σκοπιμότητα μακριά από την εκπαίδευση. Αναού του ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να διδάσκουμε την ιστορία του αυταρχισμού είναι απαραίτητο και ε, ε, ε, ως φανατική αντικομουνίστρια δεν θα σας πω εγώ το αντίθετο αλλά δεν είναι ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασχοληθεί με την εκπαίδευση κυρίως όταν εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν από την φτώχεια και ποτέ δεν βλέπουν να επιλύονται τα βασικά τους προβλήματα. Το να θέλουμε να επηρεάσουμε την έρευνα και την εκπαίδευση δεν είναι καλό μήνυμα για την ιστορική αλήθεια και αυτό το διδασκόμαστε από την ιστορία του αυταρχισμού. Και σε πολλές χώρες βλέπουμε την τάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να κινούνται προς τον ε, ε, αυταρχισμό με προπαγάνδα στα σχολεία, με διώξεις της αστυνομίας κατά των κινημάτων που είναι κατά της παγκοσμιοποίησης, όπως στην Ιταλία, στην Ελλάδα ή και στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. η ιστορία θα δείξει ε, τι σημαίνει αυταρχισμός. Κύριος Παπαδάκης, ένα λεπτό. Μιλάτε περί ολοκληρωτισμού. Ο στόχος σας προφανής, να εξισώσετε τον κομμουνισμό με το τέρας